Mes chers collègues, bonjour. Allez, on se dépêche un Καλημέρα σας, παρακαλώ να βιαστούμε λίγο. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Κοιτάω αν έχουμε ικανό αριθμό για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Κάντε πολύ θόρυβο. Est-ce Έχετε φέρει τις κάρτες σας για να ψηφίσετε. Ωραία λοιπόν, θα ξεκινήσουμε για να δούμε αν έχουμε ικανό αριθμό μελών. Ξεκινάμε λοιπόν δοκιμάζοντας τις κάρτες με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κύριε Λούγκριν, δεν δουλεύει η κάρτα μου. Ωραία. Οπότε εσείς διανατάσσεως της χειρός ή αλλάξτε ε, θέση. Really? Are you kidding me? Allez! I need to get the new one. Oh. Le groupe des Verts, on est euh, combien à voter 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 sont... votent les Verts Parce que moi, je dois voter, je crois. 1, 2, 3, 4. Ouais, je... Μετρώ τους πράσινους, άρα λοιπόν ψηφίζω κι εγώ. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας, Είμαστε όλοι εδώ λοιπόν. Τα νούμερα βγαίνουν. Λοιπόν, ξεκινάμε. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Μετροπολογίες και θα σας δώσω πάντα τα δύο τελευταία νούμερα. Θα λέω λοιπόν τα δύο τελευταία ψηφία. Το καταλάβατε? 59 θα λέω για παράδειγμα. 59 υπέρ κατά άποχες δεν είναι σαφές λοιπόν άρα λοιπόν θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία που λύγει με τα δύο ψηφία 59 ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίσατε όλοι πέρας Λοιπόν, Συν 30. Λοιπόν, να σηκώνετε και τα χέρια σας από την αρχή. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Καταπίπτει. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 08 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 ταυτόσημες 05 και 20. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 ταυτόσημες 06 και 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 04 και 18. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 09. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 καταπίπτει. Δύο ταυτόσημες που καταπίπτουν επίσης. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε κατευθείαν στην τροπολογία 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες που καταπίπτουν. 24 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτει λοιπόν. 34 υπέρ. Κατά αποχές Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για την 34 θα ψηφίσουμε μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας γιατί κάποιοι δεν σήκωσαν το χέρι τους ψηλά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συνεχίζουμε λοιπόν με την 23, με συγχωρείτε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 26, 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε αρκετές ταυτόσημες οι οποίες καταπίπτουν και περνάμε απευθείας στην 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 07 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχή εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τέσσερις 0 1, 13, 47, 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Απορρίπτεται, με συγχωρείτε. Τρεις ταυτόσημες. 02, 12 και 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 03 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεν θα γίνει συνολική πλειοψηφία. Ψηφίσαμε μόνο για τις τροπολογίες. Αχ, κύριε Ερτούκ, είχατε όρεξη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τις εργασίες μας. Ευχαριστώ πολύ, Ντομινίκ. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα τεσσάρων λεπτών, έτσι ώστε να έρθει ο κύριος Πάτρικ Κι, που είναι ο Γενικός Διευθυντής της ε, Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Αεροπλοίας στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν μέχρι να έρθει διακόπτουμε για τέσσερα λεπτά.

mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Monsieur... Σας παρακαλώ, κύριε Ερτούγκα, ξανακαθόμαστε στις θέσεις μας. Κύριε Μπάουζα ξεκινάμε. Σας παρακαλώ, κύριε Ραμόν Μπάουζα Δίας, σας παρακαλώ καθίστε και ο κύριος Ερτούγκα. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε την τεράστια χαρά να υποδεχτούμε σήμερα τον κύριο Πατρικ Κι, εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, την ΕΑΖΑ, που είναι ε, λοιπόν, ε, ο κύριος Μαρινέσκου, ειδικό γι' αυτό, εισηγητής για την έκθεση της ΕΑΖΑ, θυμάμαι ότι μείναμε μέχρι το πρωί εδώ για αυτή την έκθεση. Στην αρχή λοιπόν της νομοθετικής ε, περίοδου αποφασίσαμε να καλέσουμε εδώ τους ε, διευθυντές των τριών μεγάλων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Κί λοιπόν σήμερα θα μας παρουσιάσει την, ε, τον οργανισμό για την αεροπορία. Είχε έρθει εδώ και τον Μάρτιο, τον Απρίλιο νομίζω. Είχατε έρθει λοιπόν Κυριακή για να μας παρουσιάσετε την άποψη της ΕΑΖΑ όσον αφορά τα ατυχήματα με τα Boeing 737 MAX. Σήμερα λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να μας εξηγήσετε πού βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την υπόθεση, τι πιστεύουν οι εμπειρογνώμονες. Θα ήθελα να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση με τον Κυριακή. Σας δίνω λοιπόν Κυριακή τον λόγο για 10 λεπτά και στη συνέχεια θα κάνουμε μια συζήτηση. Μπορείτε να θέσετε λοιπόν τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις για την αεροπορία. Ευχαριστούμε Κυριακή που ήρθατε και πάλι. Έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, είναι χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι εδώ και να έχω την ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία μαζί σας. Εφόσον έχουμε νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία της σημερινής συνεδρίασης και να σας ενημερώσω πολύ σύντομα σχετικά με το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Και κατόπιν θα αναφερθώ στο 737 Max που νομίζω ότι είναι ε, πολύ ενδιαφέρον θέμα για όλους μας. Δεν ξέρω αν λειτουργεί η τεχνολογία. Όπως σας είπε η κυρία Ντελή, Ο ΕΑΣΑ δημιουργήθηκε το 2004, αλλά τον Σεπτέμβριο του 2019 είχαμε ε, έναν νέο βασικό κανονισμό που αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή σας, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκου αλλά και την κυρία Ντελή που μας υποστήριξαν και υποστήριξαν ένα διαβριμένο ρόλο για τον ΕΑΣΑ που βλέπετε στην διαφάνεια αυτή. Είμαστε η ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια της αεροπορίας, αλλά γνωρίζετε ότι η ασφάλεια της αεροπορίας περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μη οικονομική πτυχή. Έτσι, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως είναι η ασφάλεια του σκάφους, του πληρώματος, των επιβατών, των αεροδρομίων κλπ. Και με τον νέο βασικό κανονισμό, καλύπτουμε και νέα είδη αεροσκαφών όπως είναι τα τηλεκατευθυνόμενα, τα drones. Έχουμε λοιπόν έναν οργανισμό ασφαλείας στην Ευρώπη, εμάς, και με τον νέο βασικό κανονισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δέχτηκαν να ενισχύσουν το ρόλο του ΕΑΖΑ και στο περιβάλλον και θα σας ε, περιγράψω κάποιες ιδέες σχετικά με το πώς σκοπεύουμε να το πετύχουμε αυτό. Ζητώ συγγνώμη που ε, έχει τόσα πολλά πράγματα η διαφάνεια αυτή, ήθελα όμως να χωρέσω όλα τα στοιχεία σε μία διαφάνεια. Τι κάνουμε λοιπόν. Ο ΕΑΣΑ πιστοποιεί όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα εκ μέρους ε, των κρατών μελών. Τα ε, αεροσκάφη Airbus πιστοποιούνται από μας. Επίσης, προετοιμάζουμε την τεχνική νομοθεσία που υιοθετείται κατόπιν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και το περιβάλλον στον τομέα της αεροπορίας. Και κατόπιν ελέγχουμε οι κανονισμοί αυτοί να εφαρμόζονται με εναρμονισμένο τρόπο από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι, όπως ε, ίσως καταλαβαίνετε, η τεχνική εφαρμογή των κανόνων επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα του τομέα και γι' αυτό πρέπει ο ΕΑΣΑ να δημιουργεί ίσες συνθήκες ανταγωνισμού ώστε ε, να διασφαλίζουμε δίκαιο ανταγωνισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και τέλος, και αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό, καθότι η αεροπορία είναι ένας παγκόσμιος τομέας και εφόσον η Airbus εξάγει ευτυχώς το 70% των αεροσκαφών της και αντιστρόφως έχουμε αεροσκάφη Boeing, υπάρχει πολύ ισχυρός διεθνής ρόλος για τον ΝΕΑΣΑ για να προωθήσουμε και να διατηρήσουμε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο. Όσον αφορά το περιβάλλον, εμείς θέτουμε τα περιβαλλοντικά πρότυπα για τα νέα αεροσκάφη που πιστοποιούνται και υπάρχουν διάφορες προκλήσεις εδώ. Θα επανέλθω στο θέμα. Πολύ χαρακτηριστικά, όπως ίσως έχετε ακούσει, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ε, πιέζει για νέα ε, υπερηχητικά αεροσκάφη και επιστοποίησή τους ε, το 2020. Και εδώ μας ενδιαφέρουν τα πρότυπα εκπομπών και θορύβου για τα υπερηχητικά αεροσκάφη. Επίσης ε, θέλουμε να διευκολύνουμε την χρήση των ε, ε, βιώσιμων καυσίμων, να έχουμε τεχνολογίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον, όπως είναι η ηλεκτρική ή υβριδική κίνηση και να έχουμε και αντικειμενική επισκόπηση της περιβαλλοντικής απόδοσης του συστήματος αεροπορίας ή συγκεκριμένων πτυχών του. Να σας περιγράψω τις στρατηγικές μας προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία. Ο βασικός μας στόχος είναι να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις του νέου βασικού κανονισμού και ένα από τα θέματα όπου θα πρέπει να ε, εργαστούμε σκληρά είναι η καινοτομία. Έχουμε πολλά νέα ε, σκάφη, όπως είναι τα, τα drones, τα τηλεκατευθυνόμενα ή και τα αεροταξί. Επίσης, έχουμε νέα είδη καυσίμων και θα πρέπει ε, στα θέματα αυτά να πετύχουμε αποτελέσματα, ώστε να εξασφαλίσουμε οι καινοτομίε αυτές να είναι ασφαλείς. Ε, βέβαια, και η κυβερνοασφάλεια μας απασχολεί πολύ και θα πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας. Θέλουμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην ε, διεθνή σκηνή ε, να λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες των πολιτών και έγιναν πολλές συζητήσεις στο πλαίσιο του νέου βασικού κανονισμού σχετικά με τη νέα είδους σχέση ανάμεσα στις εθνικές αρχές, ε, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, και τον ΕΑΣΑ. Και αυτό είναι κάτι που προωθούμε διότι πιστεύουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες να προωθήσουμε νέους ευρωπαϊκούς παράγοντες και να έχουμε καλύτερη σχέση και καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων ε, ανάμεσα σε εμά και τις εθνικές αρχές. Όσον αφορά το περιβάλλον, ε, έχουμε δεσμευτεί να στηρίξουμε πράσινες τεχνολογίες, απαλλαγή από εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλες και θα πρέπει να εξετάσουμε το περιβαλλοντικό αντίκτυπο νέων αεροσκαφών, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον. Όλοι μιλούν για τα τηλεκατευθυνόμενα, τα drones, αλλά Συμφωνούν όλοι σχετικά με το αποδεκτό επίπεδο θορύβου από τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη στην πόλη. Ή ποιο είναι το ε, απαραίτητο επίπεδο ασφαλείας για τα αεροταξί και τα τηλεκατευθυνόμενα σκάφη σε αστικό περιβάλλον. Και τέλος, χωρίς να θέλω να πω σε πολλές λεπτομέρειες, ασχολούμαστε με το θέμα οικοσήματος, όπως για παράδειγμα όταν αγοράζετε ψυγείο, έχετε τις βαθμολογίες α, α συν, α συν συν κλπ. Εμείς θα θέλαμε να προτείνουμε κάτι παρόμοιο για τα αεροσκάφη, για τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια. Σας έκανα μια πολύ γρήγορη παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΕΑΣΑ. Επιτρέψτε μου τώρα να σας μιλήσω για το αεροσκάφος 737 MAX. Και θα προχωρήσω πολύ γρήγορα, διότι πολλά από αυτά που θα πω ήδη έχουν δημοσιευτεί στον τύπο. Δύο ατυχήματα έγιναν μέσα σε διάστημα λιγότερο από έξι μήνες και αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί στον τομέα μας. Και τα δύο ατυχήματα οφείλονταν σε παρόμοια δυσλειτουργία Το τελευταίο από τα ατυχήματα πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου του 2019 και ως αποτέλεσμα του ατυχήματος αυτού της, ε, των εθιεπικών αερογραμμών αποφασίστηκε να καθυλωθεί ο στόλος ε, στην Ευρώπη ε, και για μεταφορές προς και από την Ευρώπη. Δεν θέλω να ακρηγορήσω πάνω στο γιατί λάβαμε την απόφαση αυτή. Πιστεύουμε όμως, ε, είδαμε ότι ακολουθήθηκε η απόφαση αυτή από σχεδόν όλο τον υπόλοιπο κόσμο μετά. Και πράγματι έχετε δίκιο και ζητώ συγγνώμη. Στις 18 Μαρτίου ε, ήρθα στην Επιτροπή να σας εξηγήσω γιατί το κάναμε αυτό και να σας εξηγήσω ποιες ήταν οι πιθανές αιτίες των ατυχημάτων. Και πάλι δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά υπάρχει ένας σένσορας ε, που λέγεται angle of attack που αποφασίζει, που καθορίζει, για να το πω πολύ απλά, εάν το αεροσκάφος ε, θα ανέβει ή θα κατέβει. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε δυσλειτουργία ενό από τους δύο σένσορες. Δύο σένσορες έχει το αεροπλάνο αυτό. Και αυτή η δυσλειτουργία ε, οδήγησε το σύστημα να κατεβάσει το ρίγχος του αεροσκάφους. Και μετά την καθήλωση του στόλου, στείλαμε επιστολή στους Αμερικανούς ομολόγους μας και τους είπαμε ότι κατά τη γνώμη μας μπορεί να ε, συνεχιστεί η λειτουργία του αεροσκάφους εάν πληρούνται τέσσερις προϋποθέσεις. Καταρχάς, όλες οι τροποποιήσεις που προτείνονται από την Boeing στο σύστημα αυτό και την κινητοποίησή του να ε, εγκριθούν από τον ΕΑΣΑ. διότι έχουμε διμερή συμφωνία ασφάλειας της αεροπορίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και με την διμερή αυτή συμφωνία μπορούμε να συζητάμε, όπως άλλωστε έγινε και την αρχική πιστοποίηση του 737. Μπορούμε λοιπόν να συζητάμε τέτοια θέματα. Επιμείναμε λοιπόν ότι οποιαδήποτε τροποποίηση προταθεί από την Boeing για να αντιμετωπιστούν αυτές τις λειτουργίες θα πρέπει να εγκριθεί από τον ΕΑΣΑ. Το δεύτερο θέμα, το οποίο δεν άρεσε πολύ στους Αμερικανούς συναδέρφους μας, ήταν ότι ζητήσαμε ευρύτερη αναθεώρηση, ευρύτερη επανεξέταση ε, των συστημάτων ασφαλείας του αεροσκάφους ΜΑΞ, διότι με τη διμερή αυτή συμφωνία Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν πιστοποιήσαμε μόνοι μας, διότι είχαμε αναθέσει μερικά από αυτά στην FAA. Τρίτη προϋπόθεση ήταν η πλήρης κατανόηση ε, του τι προκάλεσε τα ατυχήματα και από τεχνικής πλευράς, αλλά και από ε, λειτουργικής πλευράς. Και τέλος, και εξίσου σημαντικό, πρέπει να φροντίσουμε για οποιαδήποτε τροποποίηση γίνει στα αεροσκάφη, θα πρέπει να λάβουν επαρκή κατάρτιση ε, τα πληρώματα. Αυτές λοιπόν ήταν οι τέσσερις προϋποθέσεις μας που ε, μεταφέραμε στους ε, Αμερικανούς τον Απρίλιο, φέτος τον Απρίλιο. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημαντικό θέμα που είναι η δική μας ε, ανεξάρτητη ε, αναθεώρηση, κατά την οποία είπαμε ότι, ωραία, στο 737 MAX Προφανώς κάποια πράγματα δεν λειτουργούσαν σωστά ε, σε συστήματα κρίσιμα για την ασφάλεια. Αλλά τι αποδειξή έχουμε ότι δεν υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου μπορεί να υπάρχουν τις λειτουργίες σε συστήματα κρίσιμα για την ασφάλεια. Γι' αυτό αποφασίσαμε να επαναπιστοποιήσουμε τα τμήματα, τα κρίσιμα για την ασφάλεια, τα οποία δεν είχαμε εξετάσει ε, στην ε, προηγούμενη ε, περίπτωση. Και λάβατε κατάλογο όλων των στοιχείων, κυρίως αναφερόμαστε στη συμπεριφορά των συστημάτων ελέγχου της πτήσης. Για να γίνει αυτό, δαπανίσαμε πολύ χρόνο και πολύ προσπάθεια. Έχουμε μία ομάδα 20 ατόμων που εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό, που συμπεριλαμβάνει μηχανούς, μηχανικούς, ε, εμπειρογνώμονες, ε, υπτάμενους μηχανικούς και Είμαστε σε στενή, σε στενή επαφή με, το, με την Boeing στο Seattle. Έχουμε 9 ώρες διαφορά όμως, οπότε μερικές φορές είναι δύσκολη η επικοινωνία. Καταφέραμε όμως να έχουμε πολύ ενεργό ψηφιακή παρουσία ε, της FAA σε όλες μας ε, τις δραστηριότητες. Ένα από τα βασικά σημεία οποιασδήποτε δραστηριότητας πιστοποίησης είναι ε, οι δοκιμαστικές πτήσεις, όπου οι πιλότοι εξετάζουν τη συμπεριφορά του αεροσκάφους και εξετάζουν εάν συμπεριφέρεται με τον τρόπο που σχεδιάστηκε να συμπεριφέρεται. Για την προετοιμασία αυτών των πτήσεων ε, έχουμε ελέγχους προσωμείωσης ε, με τους ε, πιλότους, ώστε να προετοιμαστούν για τις δοκιμαστικές πτήσεις. Είχαμε προσωμιώσεις λοιπόν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ενώ πρέπει να γίνουν οι δοκιμαστικές πτήσεις. Θα σας ενημερώσω αργότερα. Βρήκαμε σημαντικά τεχνικά θέματα. Είναι πολύ τεχνικά, γι' αυτό δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά διαπιστώσαμε κρίσιμα θέματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν προτού να μπορεί να επιστρέψει σε λειτουργία το αεροσκάφος, ιδιαίτερα όσον αφορά τον υπολογιστή ελέγχου της πτήσης και τα συστήματα ελέγχου πτήσης και την σχέση ε, αυτών μεταξύ τους, ε, καθώς ε, και τα σήματα συναγερμού που εκπέμπονται. Τον Ιούλιο επισκεφτήκαμε και την Boeing και την FAA και η Boeing έκανε κάποια πράγματα και προτείναμε και εμείς μια σειρά λύσεων που συνοψίζονται εδώ. Και πάλι πρόκειται για τεχνικά θέματα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε. Αν το θέλετε, αν είναι απαραίτητο μπορώ, αλλά θέλω ουσιαστικά να σας δείξω ότι γίνεται πολλή δουλειά πάνω στο θέμα αυτό. Από τη δική μας πλευρά γίνεται συστηματική επισκόπηση όλων των πτυχών που σχετίζονται με την ασφάλεια της πτήσης. Υπάρχουν πτυχές όπου είμαστε ικανοποιημένοι με, τα, με τις λύσεις που προτείνει η Boeing. Υπάρχουν θέματα ε, τα οποία πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω, ενώ υπάρχουν άλλα, άλλοι τομείς όπου απομένει να γίνει πολλή δουλειά. Τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την Boeing και να έχουμε πλήρη αξιολόγηση των όσων προτείνουν, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του ανθρώπινου παράγοντα. Δηλαδή, από γνωστική πλευρά, πώς μπορεί ο πιλότος ή το πλήρωμα να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα γίνουν οι δοκιμαστικές πτήσεις όταν έχουν περατωθεί επιτυχώς όλες αυτές οι δραστηριότητες και από τις δοκιμαστικές πτήσει, θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τις απαιτήσει κατάρτισης για τα πληρώματα και ιδιαίτερα θα δούμε αν χρειάζεται ε, εξάσκηση προσωμείωσης, ε, κατάρτιση σε, σε αίθουσα διδασκαλίας ε, ή άλλου τύπου κατάρτιση. Θα θυμάστε ότι στην Ευρώπη κάποια κράτη-μέλη υιοθέτησαν εθνική νομοθεσία που να απαγορεύει την είσοδο του αεροσκάφους αυτού στην, στον εναέριο τους χώρο, κάτι που δεν έγινε με πολύ συντονισμένο τρόπο. Όταν αποφασιστεί να ξεκινήσει πάλι η λειτουργία των αεροσκαφών αυτών, ε, θα πρέπει να έχουμε συντονισμένη θέση, να μην λέει ναι η μία χώρα και όχι η άλλη. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την κατάρτιση που θα χρειαστούν τα πληρώματα. Και με αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ε, πολύ βιαστικά τα είπα και ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι πολύ τεχνικό το θέμα αυτό. Ελπίζω να καταφέρατε να με παρακολουθήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ πολύ, Πατρίκ Κι, για αυτή την παρουσίαση που κάνατε, που ήταν αρκετά γενική, γιατί Ακούσαμε βέβαια και το κομβικό που είναι το αεροσκάφος ε, Boeing Max. Κύριε Μαρινέσκο, έχετε το λόγο. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας σχετικά με την εταιρεία Boeing. Έχω ένα σχόλιο το οποίο μπορεί να είναι και ερώτηση. Ένας χρόνος είναι πολύς, πολύ μεγάλη διάρκεια έχει περάσει ένας χρόνος από τα δυστυχήματα και δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι πολύς χρόνος. Τι κάνει η Boeing. Τι συμβαίνει. Γιατί κατά τη γνώμη μου πέρασε πάρα πολύς χρόνος. Και δεύτερη πολύ ανοιχτή ερώτηση. Το δυστύχημα αυτό έγινε γιατί υπήρξε πρόβλημα του αισθητήρε, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή όλα τα συστήματα backup δεν λειτουργήσαν ή δεν είχαν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν. Δεν δημιουργεί αυτό πρόβλημα αξιοπιστίας ε, της ε, σχετικής Αμερικανικής Υπηρεσίας ε, Ασφάλειας Αεροπλοείας, FAA. Ε, έχετε μια διμερή συμφωνία αμοιβαιότητας και πρέπει να τους εμπιστευόμαστε μια και δεχόμαστε τις δικές τους εγκρίσεις. Μήπως στα πλαίσια της δημερούς αυτής της συμφωνίας μπορείτε να βρείτε μια δυνατότητα να απορρίπτετε αν το σύστημα ε, κάπου χωλαίνει. Διαφορετικά, λυπάμαι που το λέω, μπορεί κανείς να φανταστεί μια επανάληψη στο μέλλον. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε ένας μόνο αισθητήρα που δυσλειτουργεί να δημιουργεί τόσο τεράστιο πρόβλημα κάτι πραγματικά πήγε λάθος. Και για το βασικό κανονισμό της ΕΑΣΑ ξέρετε πως έχετε πέντε χρόνια για να ενημερώσετε τα πάντα, όλους τους κανονισμούς και κυρίως για τη νέα προσέγγιση που βασίζεται σε αξιολόγηση κινδύνου. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των ε, πιο ελαφρών ε, σκαφών και όλων των υπολείπων. Τι γίνεται λοιπόν με το θέμα αυτό. Πού βρίσκεστε. Έχετε αρκετό προσωπικό. Έχετε αρκετά χρήματα για να φέρετε σε πέρα σε αυτή την τόσο δύσκολη δουλειά. Merci beaucoup, Ευχαριστώ πολύ κυρία Μαρινέσκου, ο κύριος Ερτούγκα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα-πρώτα για τον κύριο Κι, χαιρόμαστε που είστε εδώ σήμερα. Κύριε Κι, έχω μία ερώτηση όσον αφορά τα 737 MAX 8. Πρώτα-πρώτα ευχαριστούμε για την ενημερωσή σας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και για τις επιστολές που μου στείλατε πριν από λίγες εβδομάδες. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και ε, να δούμε τη συνεργασία σας με την FAA. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η... Ε, τι, τι νομίζετε όσον αφορά την ε, επαναπιστοποίηση. διότι οι ε, εμπειρογνώμονες στον τύπο λένε ότι δεν θα μπορέσουν να ξαναπετάξουν τα 737 MAX 8. Άλλοι πάλι λένε ότι αν λυθούν όλα τα προβλήματα και ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού, τότε και πάλι θα επανέλθουν σε λειτουργία. Η δική μου άποψη προσωπικά είναι ότι πραγματικά θα δίσταζα στο μέλλον να πετάξω με ένα 737. Το θέμα είναι ψυχολογικό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αξιολόγηση της επαναπιστοποίησης, το θέμα που θα ήθελα να σας θέσω, και επίσης όσον αφορά τις ε, απαιτήσει κατάρτισης, ε, αν θα πρέπει να ε, θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος ε, της ε, πιστοποίησης για το σκάφος και πιο συγκεκριμένα για την κατάρτιση και τις απαιτήσει για αυτήν. Θα είναι δυνατόν να είναι οι ίδιες οι απαιτήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ, όπως γίνεται και για τις ε, τεχνικές. Ευχαριστώ κύριε Ερτούγκ. Ο κύριος Μπαουζαντίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Κι και για το ότι είναι εδώ, αλλά και για τη διάδοση πολύ λεπτομερείς εξηγήσει για την περίπτωση του Boeing 737 MAX. Έχω κανένα δύο ερωτήσεις και δεν θα ήθελα να χάσω την ευκαιρία, μια και είστε και εσείς εδώ, γιατί με ενδιαφέρει πολύ το τι θα γίνει στο μέλλον και έχουμε και το Brexit. Νομίζω πως είναι σημαντικό να τονίσουμε πως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αποτελεσματική και συντονισμένη στις προσπάθειες που θα, που θα κάνει για να αποφύγει τις πολύ βλαβερές συνέπειες της απόσυρσης ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από την σχετική νομοθεσία για την αεροπλία. Και θα ήθελα επίσης να σεβαστούμε τους κανονισμούς της προηγούμενης θητείας και κυρίως για τα contingency plans, τα σχέδια ασφαλείας, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλείς αερομεταφορές και να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε την αμοιβαιότητα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα ήθελα να μου απαντήσετε λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον πλαίσιο. Ποιες είναι οι σχέσεις ε, της δικής σας υπηρεσίας με την Ομόσπονδη αντίστοιχη η υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών με την αμοιβαία αναγνώριση προτύπων ασφαλείας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε για το πώς η υπηρεσία επενεύει στην ε, ανάλυση των δυστυχημάτων πριν και μετά και ποιες, ποιοι ήταν οι παράγοντες ε, με τους οποίους ε, ασχολήθηκαν οι δικοί σας εμπειρογνώμονες εσωτερικοί και εξωτερικοί και τι σημαίνει αυτό για την περαιτέρω εκπαίδευση των πληρωμάτων έτσι ώστε να αποφύγουμε ίδια δυστυχήματα στο μέλλον. Η FAA τι κάνει σχετικά. Ποιος θα είναι ο ρόλος σας για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου μας σε μια αγορά που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Βλέπουμε τι γίνεται όχι μόνο με τους Αμερικάνους αλλά και με τους Κινέζους. Τι κάνετε εσείς για να προωθήσετε τη δική μας συνεισφορά στη μείωση των εκπομπών έτσι ώστε να μην γίνει ο κλάδος μας μη ανταγωνιστικός. Και βέβαια θα σας ξαναευχαριστήσω για τις εξηγήσει που μας δώσατε για τα όσα συνέβησαν με τα δυστυχήματα του Boeing 737 MAX ήταν εξαιρετικές και είχα πάρα πολλές ερωτήσεις και τις απαντήσατε εσείς πριν προλάβω να τις κάνω. Μιλήσατε με πολλές λεπτομέρειες και χαίρομαι γιατί απαντήσατε πολύ συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόφ. Ευχαριστώ. Έχω κι εγώ μια ερώτηση για το τι κάνει η FAA που είναι η αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ομόσπονδη, γιατί είναι προφανές ότι οι τραγωδίες που συνέβησαν με τα Boeing 737 MAX είναι εξαιρετικά ζημιογόνες για το κύρος της FAA. Και είναι και ένα παράδειγμα ε, θεσμικής ε, παρέτησης ε, Κάποιε ομόσπονδες υπηρεσίας. Εσείς λοιπόν αυτή τη στιγμή τους κοιτάτε κατάματα. Και τι αισθάνεστε, εκπροσωπούν τον κλάδο ή τον κόσμο που ταξιδεύει. Γιατί για μένα είναι προφανώς η FAA είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ ευάλωτη θέση, τους πλήγωσε πολύ. Και δεν ξέρω αν αυτό ε, επηρεάζει σας; και το πώς αναγνωρίζετε εσείς ε, τα όσα έχουν κάνει και πώς βλέπετε εσείς στο μέλλον να διαμορφώνετε οι σχέση σας με αυτούς. Η άλλη μου ερώτηση έχει να κάνει με την ε, αεροπλοεία και κυρίως με την ηχορύπανση στα αεροδρόμια. Την επόμενη δεκαετία πιστεύω πως ο ήχος θα αυξηθεί, η ηχορύπανση μάλλον, και δεν ξέρω τι αρμοδιότητες έχετε εσείς για να περιορίσετε ή να ελέγξετε ε, την ηχορύπανση που προέρχεται γενικότερα από την αεροπλοεία. Γνωρίζουμε ότι είναι επιζήμια η ηχορύπανση για την ανθρώπινη υγεία και δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι έχετε όλες τις αρμοδιότητες που χρειάζονται για να ελέγξετε και να μειώσετε την ηχορύπανση από τα αεροσκάφη και από τα αεροδρόμια και κυρίως εν ώψη των πιέσεων που αντιμετωπίζεται από τις ΗΠΑ και από τις αρχές των ΗΠΑ. κυρία Λεσοντέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Διευθυντή, το θέμα της ασφάλειας ε, που θίξατε συνδέεται πάρα πολύ στενά με τις συνθήκες εργασίας ε, για τους εργαζόμενους στον κλάδο. Και η δική μας στρατηγική ε, για την αεροπλοεία λαμβάνει υπόψη την κοινωνική προστασία. Και το Μάρτιο πέρσι καταγγείλαμε μια κατάσταση εργασιακή απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας. Η έκθεση Ρικάρντο που ανέφερε η Επιτροπή στην αγορά έχουμε πολλά προβλήματα. Απόσπαση εργαζομένων, ε, συμβασιούχοι, ε, σύντομες συμβάσεις, έμεση απασχόληση και καθεστώτα ε, διαφορετικά για πληρώματα από τρίτες χώρες. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά επίμαχα και έχει να κάνει με την απόσπαση που χαρακτηρίζει τις συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων. Επειδή λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε με τη δική σας ε, υπηρεσία για να εξασφαλίσουμε πως η ασφάλεια των αεροπορικών εταιριών λαμβάνει υπόψη όλες τις κατηγορίες εργαζομένων και όλα τα καθιστώτα υπό τα οποία προσλαμβάνονται, θέλω να μου εξασφαλίσετε ε, πως η ασφάλεια λαμβάνεται υπόψη δεόντως ως πρώτη προτεραιότητα, αλλά και οι εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων επίσης εξετάζονται από εσάς. Σας ευχαριστώ. Κυρία Νταλή. Ε, um, Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω τον ρόλο που παίξατε στα Boeing 737, αλλά νομίζω ότι τα ατυχήματα αυτά μας δείχνουν και κάποιες αδυναμίες σε επίπεδο εργάνωσης όσον αφορά την εφαρμογή. Είπατε ότι το 2000, είχατε πει μάλλον το 2016 ότι η Boeing είχε δεχτεί κατάρτιση του πληρώματος ανάλογη, όμως αυτή η κατάρτιση δεν έλαβε ποτέ χώρα. Σήμερα λοιπόν μας λέτε ότι η Boeing σας διαβεβαιώνει και πάλι ότι τώρα θα καταρτήσει τα πληρώματά της. Ε, γιατί θα αλλάξουν τα πράγματα, γιατί πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Νομίζω ότι σωστά είπαν οι συνάδελφοι για την FAA ότι δεν έχουμε εκεί επιρροή. Και αναρωτιέμαι, ιδίω όσον αφορά ανάλογα προβλήματα, όσον αφορά τα συστήματα ε, που είναι κρίσιμα για την ασφάλεια. Πώς θα μπορούσατε να μας εγγυηθείτε εσείς ότι η πιστοποίηση των Airbus θα είναι επαρκής. Ποιες οι διασφαλίσεις μπορείτε να μας δώσετε. Νομίζω ότι δεν μπορέσαμε να... Ε, μάλλον, μπορέσατε να εντοπίσετε κάποια προβλήματα με τα 737, αλλά δεν μπορέσατε να επιβάλλετε μέτρα. Τι, ε, λοιπόν, μπορούμε να αντλήσουμε από όλα αυτά. Επίσης, τον Μάρτιο μας είπατε όσον αφορά τον ε, περιορισμό ε, χώρου, ε, χρόνου πτήσης για τις νυχτερινές πτήσεις. Οι, οι νυχτερινές πτήσεις βεβαίως διαταράσσουν το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου και εδώ τίθενται και θέματα όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατών. Τι προτίθεστε λοιπόν να κάνετε γι' αυτό και πότε θα προτείνετε αλλαγές όσον αφορά τον προγραμματισμό των ε, πτήσεων στην Ευρώπη, κυρίως όσον αφορά τις νυχτερινές πτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Σκότ. Ευχαριστώ πολύ. Είχα πολλές ερωτήσεις που τις, ε, απάντησαν, τις έκαναν μάλλον ήδη οι συνάδελφοι. Θα πρέπει όμως να τις απαντήσετε. Αυτό που με ανησυχεί εμένα ιδιαίτερα, με βάση την ενημέρωση που μας κάνατε, είναι αυτές οι διαδρομές ε, πτήσεων που μου φαίνονται παρόμοιες. Επίσης το θέμα της έλλειψης καταρτήσεων για τους πιλότους, για το προσωπικό. Πολλά είναι τα θέματα λοιπόν που πρέπει να απαντήσετε. Αλλά εδώ πρόκειται για ένα ανθρώπινο λάθος, για ένα λάθος μηχανής. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν και περιμένουμε απαντήσεις. Η συγκεκριμένη ερώτηση που θέλω εγώ να θέσω είναι η εξή. Πολλοί ε, ε, συνάδελφοι μίλησαν για το Brexit. Σε περίπτωση λοιπόν μη συμφωνίας, ανάλογα με το τι θα γίνει ε, την 31η Οκτωβρίου, ποιο θα είναι το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου εντός του οργανισμού σας και ποιες θα είναι οι ε, επιπτώσεις για τις διεθνείς πτήσεις εντός και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ. Κύριε Ετιάν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κύριε Κάι, έχω μία ερώτηση σχετικά με το θέμα του Boeing και συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα. Για μένα είναι σαφές ότι η ασφάλεια θα πρέπει να προέχει και δεν θα πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στο θέμα αυτό. Ε, δεν εξαρτάται λοιπόν από εσά το πότε θα έχει απαντήσει η Boeing σε όλε τι ερωτήσει και πότε ε, θα έχει εκπληρώσει όλε σα τι επιθυμίε, αλλά μια εκτίμηση θα ήθελα από εσά. Κατά τη γνώμη σα, ε, πόσο θα διαρκέσει μέχρι τα 400 καθυλωμένα αεροσκάφη να μπορούν να ξαναπετάξουν και τα 300 που έχουν ε, κατασκευαστεί, που δεν έχουν πετάξει ακόμα όμως, να μπορούν να απογειωθούν και η κατάρτιση των πληρωμάτων και όλα αυτά, πόσο καιρό θα διαρκέσουν. Και μία πιο γενική ερώτηση. Όλοι αγωνιζόμαστε ώστε να γίνει πιο πράσινη, πιο οικολογική η αεροπορία και πιο βιώσιμη. Για μένα λοιπόν τίθεται το ερώτημα. Έχουμε προβλήματα με ε, τις μπαταρίες, τους συσσωρευτές ε, στα αεροσκάφη και λόγω βάρους και λόγω ασφαλείας. Πότε πιστεύετε ότι τα βιοκαύσιμα θα μπορούν ε, να συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ώστε να χρησιμοποιούμε όχι μόνο υβριδικές και ηλεκτρικές τεχνολογίες, αλλά να ε, έχουμε και ε, βιολογικά καύσιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε η κυρία Δήλαου. Με συγχωρείτε δεν σας είδα. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Η μία όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια. Και στην αεροπλοεία, λοιπόν, το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την ασφάλεια των ευρωπαϊκών προτύπων, αλλά και τα διεθνή πρότυπα. Οι ευρωπαϊκές αρχές λοιπόν και η συνεργασία τους είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτόν τον τομέα προκειμένου να διασφαλίσουμε ε, λοιπόν την ασφάλεια. Υπάρχει και ο σχετικός ευρωπαϊκός ε, κανονισμός. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ο ΕΑΣΑ όσον αφορά την ενέργεια ασφάλεια, τι μπορεί να κάνει για την κύβερνο ασφάλεια και πώς μπορούν ε, οι οργανισμοί να συνεργαστούν μεταξύ τους και τι μπορούν να κάνουν και ε, σε επίπεδο χρηματοδοτικό, ούτως ώστε να υπάρχει ομογενοποίηση όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους. Επίσης, ε, τι μπορούμε να κάνουμε μέσω πρόθεσμα για προστασία κατά της τρομοκρατίας ε, και για να προστατεύσουμε την πολιτική αεροπορία στην Ευρώπη. Επίσης, όσον αφορά τον εναέριο χώρο, ο ΕΑΣΑ έχει νέες αρμοδιότητες όσον αφορά τα drones. Έχει πλέον και εκτελεστικές δυνατότητες. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του εναέριου χώρου όσον αφορά τα drones. Από τη μια ακούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν, ότι να είναι οι ίδιοι οι πάροχοι που να διασφαλίζουν την διαχείριση. Όμως δεν μπορούμε να ξεχνάμε και το θέμα της ασφάλεια, που είναι πολύ σημαντικό. Αναρωτιόμαστε λοιπόν εάν οι πάροχοι στην αγορά μπορούν να είναι πραγματικά αξιόπιστοι ω προς αυτό, διαφορετικά εάν θα έπρεπε όσον αφορά λοιπόν την ασφάλεια να αναθέσουμε αλλού το θέμα. Επίσης υπάρχει το θέμα του θορύβου, κυρίως όσον αφορά τα αεροδρόμια, κυρίως κατά την απογείωση και την προσγείωση. Ο ΕΑΣΑ λοιπόν έχει, ε, προβλέπει και στο μέλλον κάποιες ε, ε, πρωτοβουλίες ως προς αυτό, προκειμένου να προστατευτεί και ο τοπικός πληθυσμός. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκυζέκια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρική, σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Ε, πράγματι, η ε, οι συνάδελφοι ρώτησαν σχεδόν τα πάντα. Είναι δύσκολο να βρω μια ερώτηση. Έχω μια ερώτηση όμω που έχει να κάνει με την αρχική σα δήλωση, τα μελλοντικά καθήκοντα του ΕΑΖΑ. Είπατε ότι θέλετε νέου είδου σχέση με τι ε, εθνικέ ε, αρχέ αεροπορία και τον σχετικό βιομηχανικό τομέα. Θα ήθελα λοιπόν εδώ συγκεκριμένη απάντηση. Τι ακριβώς θέλετε να αλλάξετε στις σχέσεις αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Κόβαρικα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω ένα από τα θέματα που γύραν και οι προηγούμενοι ομιλητές. όσον αφορά κάποια θέματα που αναφέρατε για τον νέο βασικό κανονισμό για τα drones. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο ποιες είναι οι προσδοκίες σας όσον αφορά την νομοθεσία κυρίως όσον αφορά θέματα ε, ε, παρενόχλησης της κυκλοφορίας που σημειώθηκαν στο παρελθόν, ε, στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης έχουν συμβεί, ίσως και στο Χήθρο. Ίσως μπορείτε επίσης να μας πείτε περισσότερα για τις ε, απαιτήσεις ε, καταχώρησης. Επίσης δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό το θέμα. Ο ΕΑΣΑ συνεργάζεται και με άλλες αρχές, όπως αυτές του Καναδά, για παράδειγμα, όσον αφορά τα drones. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. Και μια άλλη ερώτηση, κάπως ιδιαίτερη. Όσον αφορά ένα συγκεκριμένο συμβάν, ε, μια συγκεκριμένη πτήση που πήγε από τις ε, στις 27 Αυγούστου ένα, ήταν ένα Boeing 737 το οποίο πετούσε επί δύο ώρες χρησιμοποιώντας μόνο ένα κινητήρα. Έκανε μια δήλωση ο ΕΑΣΑ μετά από αυτό το συμβάν και ε, εδώ παραθέτω έλεγε ότι είχε ότι θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση το... Ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να πηγαίνει σε, ε, να παρακάμπτε την πτήση σε άλλο αεροδρόμιο. Όμω εδώ το θέμα παραμένει: υπήρχε ένα μόνο κινητήρα, πήγε έτσι στον τελικό του προορισμό το αεροπλάνο και ε, σήμερα γίνεται μια έρευνα από τις αρμόδιες αρχές και άλλοι έχουν εκφράσει ανησυχίες όσον αφορά το συμβόν αυτό, κυρίως διότι το πλήρωμα λέγεται ότι δεν πληροφόρησε για το πρόβλημα αυτό, τις αρμόδιες αρχές. Σκοπεύετε να κάνετε μια έρευνα ως ΕΑΣΑ για αυτό το συμβάν. Θεωρείται από αρκετούς εμπειρογνώμους ότι είναι πολύ σημαντικό. Και πιο γενικά, νομίζετε ότι όσον αφορά τις ε, απαιτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύετε ότι είναι αρκετά αυστηρές σε σχέση με αυτές της FAA, ε, όσον αφορά τέτοιες περιπτώσεις. Ε? Δηλαδή ότι η FAA απαιτεί σε αυτές τις περιπτώσεις να προσγειώνεται το αεροπλάνο. Ευχαριστώ. Πρέπει να επιταχύνουμε λίγο, γιατί υπάρχουν πολλοί ομιλητές που πρέπει να πάρουν το λόγο. Η κυρία Άννα Ντεβαγνέ. Κυρία Πρόεδρε, Κι, εμείς ως πράσινοι ενδιαφερόμαστε κυρίως για τον οικολογικό μετασχηματισμό και στον τομέα της αεροπλοείας. Μας είπατε ότι κατανοείτε ε, βεβαίως ότι πρέπει να ε, κάνουμε κάτι για το κλίμα, για την κλιματική αλλαγή, αλλά ε, παράλληλα να έχουμε και αεροπορική ασφάλεια. Αυτή είναι η εντολή σας. Ποια μέσα έχετε ή τι χρειάζεστε ως οργανισμός για να μπορέσετε να εφαρμόσετε την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και του διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, όσον αφορά τα τέλη προσγείωσης, ε, πώς μπορούμε να τη μεταλλευτούμε για το περιβάλλον. Στο αεροδρόμιο στην ε, Στουτγάρδη, ξέρω ότι εφαρμόζεται, αλλά σε διεθνές επίπεδο, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διεθνή εμπειρογνωμοσύνη, πώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε εσείς ως οργανισμός, ε, για να, καταλάβουμε, να καταλάβετε καλύτερα ποιες είναι οι άλλες ανάγκες, για παράδειγμα τέλη επί της κυροζήνης κτλ. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Merci beaucoup. Schulz. Ευχαριστώ κύριε Σούλς. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Δύο-τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις έχω σχετικά με τα ατυχήματα που περιγράψετε με τα αεροσκάφη 737 MAX. Ε, είναι γνωστά αυτά. Υπάρχουν όμως αναφορές στα ε, στον τύπο από πιλότους που ε, είπαν ότι υπήρξαν ε, προβλήματα πριν τα ατυχήματα τα οποία ανέφεραν. Τι έγινε λοιπόν και δεύτερον. Πράγματι, στην αρχική φάση είχε κανείς μόλις μερικά δευτερόλεπτα να κλείσει κανείς αυτό το σύστημα. Μήπως ε, υπήρχε πρόβλημα πληρωμάτων άπειρων. Μήπως έχουν αποφευθεί δηλαδή ατυχήματα από πιο έμπειρα πληρώματα. Και τρίτον υπήρξαν προβλήματα τέτοια που δεν οδήγησαν σε σύγκρουση του αεροπλάνου, αλλά όπου ε, ο σωστός χειρισμός από το πλήρωμα μπόρεσε να προλάβει ε, κάποιο ατύχημα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρόμαστε, Πάτρικ, που είσαι μαζί μας. Έχω μία ερώτηση όσον αφορά το Boeing Max. Νομίζω ότι κανένας δεν είπε το αντίθετο. Η FAA είχε εμπιστευτεί στον ε, τον ίδιο τον κατασκευαστή την πιστοποίηση, την είχε αναθέσει. Κυρίως όσον αφορά αυτόν τον μηχανισμό διόρθωσης που έχει να κάνει την ισορροπία του αεροσκάφους. Ο ΕΑΣΑ, λοιπόν, όσον αφορά την αυτοπιστοποίηση του κλάδου, δηλαδή κάνει την ανάθεση αυτή στους κατασκευαστές, και όσον αφορά αυτή την αυτοπιστοποίηση, Μπορούμε να αμφισβητήσουμε λοιπόν αυτή την διαδικασία πιστοποίησης εκ μέρους της FAA. Υπήρξε, υπήρχαν διεθνή, υπήρξαν διεθνείς αντιδράσεις όσον αφορά την διαδικασία της αυτοπιστοποίησης. Και μια άλλη ερώτηση. Ο ΕΑΣΑ έχει ενισχυθεί εδώ και δύο-τρία χρόνια όσον αφορά την κυβερνασφάλεια είναι αλήθεια ή αναθέτει και σε άλλους οργανισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κέ για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Τονίσατε ποιος είναι ο ρόλος της ΕΑΣΑ για την ασφάλεια και μιλήσατε κυρίως για τα τεχνικά σημεία. Όπως είπε και κάποια άλλη συνάδελφος, δεν μιλήσατε καθόλου για την κοινωνική διάσταση που πολλές φορές δημιουργούν κινδύνους. Κάτι πολύ κρίσιμο. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συμβάσεις που έχουν οι πιλότοι, με μηδενικές ώρες, με ε, μπλοκάκια, ε, θέματα τα οποία κάνουν το ταξίδι ολόκληρο επικίνδυνο. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα της κόπωσης, όχι αρκετές ώρες ξεκούρασης, υποχρέωση να δουλέψεις ε, όσο ασθενής. Είναι δηλαδή αυτές οι ευάλωτες συνθήκες εργασίας που δεν ωφελούν την ασφάλεια των πτήσεων. Και δεν ξέρω αν έχετε λάβει κάποια μέτρα για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φερέιρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον εκτελεστικό διευθυντή της υπηρεσίας και να σας κάνω τις εξής δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, επιπτώσεις για το περιβάλλον. Δεν μιλώ μόνο για τα καινούργια αεροσκάφη, αλλά και για αυτά τα συμβατικά τα οποία πετάνε σήμερα, όπως είπατε και εσείς, η χορύπανση και οι είναι όλο και περισσότερες. Και τονίσατε πως υπάρχει ανάγκη να θεσπίσουμε αυστηρούς κανόνες για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία. Έχουμε μία μελέτη του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας που έχει να κάνει με τα μικροσωματίδια και τις εκπομπές αυτών στον ε, τομέα της αεροπλοείας. Έχουμε κάποια ανώτατα όρια ε, για τα μικροσωματίδια ε, αλλά δεν έχουμε για τα υπερβολικά μικρά μικροσωματίδια κάτω από συγκεκριμένα μεγέθη για τα αναπνευστικά και νευρολογικά προβλήματα που ενδεχομένως μπορούν να προκαλέσουν. Και σύμφωνα με τη μελέτη αυτές, οι ανώτατες τιμές ε, είναι εξαιρετικά υψηλές γύρω από τα αεροδρόμια, για παράδειγμα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν θα κάνετε κάτι σχετικό για να το αντιμετωπίσετε. Επίσης, για το θέμα της χορύπανσης. Είναι ξεκάθαρη η συνέπεια που έχει για την ανθρώπινη υγεία και εκεί νομίζω είναι απερίφραστη και η νομοθεσία. Τώρα, περνάμε στο θέμα της εταιρεία Airbus και το νέο σκάφος το οποίο ξεκίνησε ε, κυκλοφόρησε στην αγορά πέρυσι που λοιπόν, το Α330. Ξέρετε κι εσείς πως είχαμε κάποια ε, κάποια ζητήματα, μία ε, δυσφορία των επιβατών ε, και του πληρώματος μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, ναυτία, εμετό, λιποθυμία, ε, απώλειες θύσεων, Αυτά σας τα έχουν κοινοποιήσει? Νομίζω πως ναι. και πιστεύω πως το θέμα αυτό θα πρέπει να το εξετάσετε. Αν δεν, αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποια λάδια μπήκανε στον ε, κινητήρα υψηλή συμπίεση και από εκεί είχαμε διάχυση στην καμπίνα. Ε, το έχετε συζητήσει με τον κατασκευαστή. Επόμενη. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς και τον κύριο Κή για τις εξηγήσεις που έδωσε. Να σας πω πως είμαστε πολύ σημαντικοί από το 2019 και μετά. Η υπηρεσία σας έχει περισσότερες αρμοδιότητες γιατί όλες αυτές οι υπηρεσίες ε, μεγαλώνουν ε, μέσω των διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν, προκλήσεων, συγκρούσεων κτλ. Ήθελα να σας ρωτήσω τα εξή πώς θα ενισχύσουμε την διεθνής, την διεθνή μας ε, θέση. Έχετε κάποια στρατηγική ε, για το θέμα αυτό και μιλώντας για την ε, πράσινη τεχνολογία. Έχουμε προβλήματα με την αυτοκινητοβιομηχανία και με τα ηλεκτρικά οχήματα σε επίπεδο αυτοκινήτων. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι όταν μιλάμε για τα αεροσκάφια χρειαζόμαστε μεγαλύτερη περισσότερο ενδιαφέρουν από τη σχετική βιομηχανία. Πιστεύετε πως οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί στηρίζουν επαρκώς την αεροναυπηγική βιομηχανία έτσι ώστε να ξεκινήσει η μελέτη για την εφαρμογή νέων βιώσιμων τεχνολογιών, ηλεκτροκίνησης κτλ. Τέλος, επειδή χρειαζόμαστε ένα καινούριο πλαίσιο για τα νέα οχήματα, μιλάμε για μη επανδρομένα αεροσκάφη, εσείς είπατε πως δεν έχουμε ακόμα τη σχετική συμφωνία, ούτε καν για τα επίπεδα ηχορήχανσης. Όταν πια θα έχουμε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τα αεροταξί, έχουμε μη επανδρομένα εξαιρετικά εξελιγμένα που θα αναλαμβάνουν καθήκοντα που σήμερα δεν ασκούν τι θα γίνει με τις σχέσεις μας με άλλες χώρες. Και επίση, όταν έχουμε τόσο δυναμικές βιομηχανίες στην Ευρώπη που κατασκευάζουν αυτά τα ντρόουν, ε, τι θα κάνετε, πώς αξιολογείτε εσείς το μέλλον και τι θα έπρεπε εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ κυρία Μπιλπάου. Κυρία Νατικάλβο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Κι. Το καλοκαίρι διάβασα ένα άρθρο στις εφημερίδες μάλλον εγώ το έγραψα, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στα αεροπλάνα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι πολλοί επιβάτες έχουν κακή συμπεριφορά μέσα στα, αεροδρόμια, μέσα στα αεροπλάνα. Δεν φέρονται καλά. Και αυτό δημιουργεί ιδιαίτερο άγχος στους άλλους επιβάτες. Μερικοί μάλιστα επιβάτες είναι και βίαιοι στη συμπεριφορά τους. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε γι' αυτό. Ε, έχετε εξετάσει το θέμα ως ΕΑΣΑ και προτίθεστε να κάνετε κάτι για να το βάλετε κάτι ε, στο θεματολόγιο των διαφορετικών ε, αερογραμμών ε, εταιριών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ δύο-τρεις ερωτήσεις για σας, Κυριακή. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ε, όλα αυτά που μας είπατε, για την ανάλυση σας, αλλά υπάρχει κάτι ε, το οποίο δεν πρέπει να συγχαίουμε με όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορούμε να γενικεύουμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε ε, την ορολογιακή βόμβα του κλίματος στον πλανήτη. Όταν βλέπουμε τον, τα δάση του Αμαζονίου σήμερα, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η αεροπλοεία είναι σήμερα ε, το 3% λοιπόν των παγκόσμιων εκπομπών αερίων ε, του θερμοκηπίου και είναι ο μόνος τομέας που δεν τους μειώνει. Έχουμε όλο και περισσότερα αεροπλάνα τα τελευταία χρόνια και ε, σήμερα πάνω από το 21% λοιπόν των μεταφορών είναι εναέριες. Δεν φτάνουν ούτε τρεις πλανήτες γι' αυτό. Η κατάστασή μας λοιπόν είναι δεινή. Η πρώτη με ερώτηση λοιπόν είναι πολύ απλή. Ξέρω ότι ο ΕΑΣΑ προβληματίζεται εδώ και πολλά χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά όταν σας ακούω να λέτε ότι ναι, ε, θα βρούμε θετικά καύσιμα για το περιβάλλον, εγώ δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα καύσιμα. Τι θα πει αυτό. Υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο για την αεροπλοεία που θα μας οδηγήσει, που θα μας βγάλει μάλλον από το φινικέλαιο που εμείς οι ίδιοι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε αποκλείσει, που έχουμε πει ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθεί από το 2021. Τίθεται όμως πάντα το θέμα. Φινικέλαιο σημαίνει αποδάσωση. Και σήμερα δεν μπορούμε πλέον, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ε, καταστρέψουμε δάση επιπλέον. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα περίφημα θετικά καύσιμα. Επίσης, ποια άλλη είναι οι τομή στους οποίους μπορούμε να εργαστούμε. Για παράδειγμα, δεν σας άκουσα να λέτε κάτι, νομίζω, πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις ε, εναέριες ροές στους εθέρες. Δεν θα επανέλθω στο θέμα του θορύβου, της ηχορύπανσης, μιλήσαμε ήδη αρκετά. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάπως περισσότερο τι εννοείτε με το οικολογικό σήμα, το ε, eco-label, Όσον αφορά τα αεροπλάνα, όπως μας είπατε, πώς λοιπόν θα υπολογίζετε τις εκπομπές άνθρακα στον τομέα αυτό. Και κάτι άλλο, για μένα σημαντικό και που διαπιστώσαμε σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στις German Wings, υπάρχουν σήμερα πιλότε οι οποίοι είναι ιδιαίτερα, έχουν ιδιαίτερο άγχος και Βεβαίω, σε αυτό το δραματικό επεισόδιο τη German Wings είχατε κάνει μια σημαντική σύσταση, δηλαδή να μην αφήνουμε μόνου στην καμπίνα, στο πιλότηριο του πιλότου, αλλά να υπάρχει πάντα κάποιο από το υπτάμενο πλήρωμα που να είναι μαζί του. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο. Σήμερα λοιπόν, έχετε κάποια νέα στοιχεία όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Τι γίνεται λοιπόν στο πιλωτήριο ούτως ώστε να ε, διευκολύνουμε την κατάσταση για τους πιλότους. Και όσον αφορά το θέμα του Brexit, είναι ένα πραγματικό θέμα, ρεαλιστικό θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν, είναι χρόνια τώρα που θέλουμε να κάνουμε κάτι, γιατί με το θέμα του Brexit Έχουμε βεβαίω επανατίθεται το θέμα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Τι σκέφτεστε λοιπόν, πώς θα προλάβετε την κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν βρετανικό κεφαλαίο ακόμα και αν ε, ε, υπάρχει συμφωνία από τη στιγμή που αυτή δεν θα εφαρμόζεται. Τι προτίθεστε να κάνετε. Σκέφτομαι κυρίως την Ισπανία που εξαρτάται ιδιαίτερα από βρετανικές αεροπορικές εταιρείες. Επίσης, δεν μιλήσαμε αρκετά για την ψηφιοποίηση, που είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Και εγώ όσον αφορά την ψηφιοποίηση έχω ένα σημαντικό πρόβλημα. Μιλάμε για drones. Και εδώ νομίζω ότι δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι όσον αφορά την άδεια για τα drones. Μας μιλάτε για τα αεροταξί και την ψηφιοποίηση, εδώ τίθεται το θέμα των δεδομένων. Και κανένας δεν το λέει ξεκάθαρα. Όμως ξέρουμε ότι τα θέματα, το θέμα των δεδομένων θα είναι το τεράστιο θέμα του αύριο. Και πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Ρίκε, ε, όσον αφορά την ε, ε ομογενοποίηση, την, ε, όσον αφορά την αδειοδότηση αυτών των συσκευών. Μήπως στο μέλλον θα μπορέσουμε να σας δώσουμε, ναι, κάποια χρηματοδοτικά μέσα, διότι ξέρουμε ότι ο προπολογισμό σας δεν έχει αυτές τις δυνατότητες. Τι μπορούμε να κάνουμε. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ε, ομαδοποιώντας τις ερωτήσεις ανά θέμα. Καταρχάς, Brexit. Ο ΕΑΣΑ δεν έχει εντολή ή κάποιο εργαλείο στην αρμοδιότητά του για να εξετάσει τα δικαιώματα κυκλοφορίας ή την ιδιοκτησία των αεροπορικών εταιριών. Δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω στο θέμα αυτό. Είμαστε αρμόδιοι για την εφαρμογή ενιαίων ε, προτύπων ασφαλείας για όλα τα αεροσκάφη που πετούν εντός της Ευρώπης και προς την Ευρώπη. και μπορώ να σας πω ότι για όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια μπορούμε να διαχειριστούμε την ε, κατάσταση μετά το Brexit. Φυσικά θα υπάρξουν κάποιες πιο εύκολες, πιο δύσκολες λύσεις, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. για να δώσουμε άδεια σε βρετανικές εταιρείες που θα παρέχουν υπηρεσίες σε ε, ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ε, συνήθως μιλάμε για συντήρηση. Για παράδειγμα, μια πτήση της Air France προς το Λονδίνο μπορεί να λάβει κάποιες υπηρεσίες από μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που θα πρέπει να έχει επιστοποιηθεί από εμά. Αυτό λοιπόν έχουμε κάνει για την κατάρτιση, για την συντήρηση και για άλλες υπηρεσίες. Από 800 βρετανικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, νομίζω ότι έχουμε επιστοποιήσει τις 700. Επίσης, έχουμε συνεργαστεί με τον βιομηχανικό τομέα όσον αφορά τους προμηθευτές ε, για την Airbus, για παράδειγμα, ώστε να αποφύγουμε ε, τις λειτουργίες ε, διαταράξεις ε, όσον αφορά την προμήθεια και τέτοια. Βέβαια, θέμα θέματα επιμελητίας είναι άλλο θέμα, αλλά πιστεύουμε ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να διασφαλίσουμε από τη δική μας ε, πλευρά να έχουμε όσο γίνεται πιο ομαλή λειτουργία μετά το Brexit. Μπορεί να υπάρξουν πράγματα που δεν έχουμε προβλέψει, αλλά νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά προετοιμασμένοι για την κατάσταση που θα επικρατήσει. Να απαντήσω σε μια από τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Σε περίπτωση ε, ασύντακτου Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει τρίτη χώρα. Δεν θα πια, δεν θα είναι πια μέλη του ΕΑΣΑ. και όλε οι επιχειρήσει, όλοι οι οικονομικοί φορεί που θέλουν να λειτουργήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περάσουν από πιστοποίηση ε, τρίτης χώρας ε, στον ΕΑΣΑ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε, είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Σε περίπτωση πάντως Brexit χωρίς ε, συμφωνία... Δηλαδή, αυτό που λέτε είναι ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει χωρίς συμφωνία, τότε θα είναι υποχρεωμένο να δημιουργήσει το δικό του οργανισμό και ότι η Ευρώπη δηλαδή μπορεί πλέον να ελέγξει την ασφάλεια και την ασφάλεια των επιβατών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Α, αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, να το καταλάβουμε καλά. <laughs> Euh, Όντως, Το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να προσλαμβάνει το απαραίτητο προσωπικό για να δημιουργήσει την τεχνική ικανότητα και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα τμήμα ε, του ε, σχεδίου που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή το Recovery Plan. Έχουμε κάποιες χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρώπης, με τις οποίες έχουμε εξαιρετικά ισχυρή ε, εταιρική σχέση, αλλά αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο απάντηση θα δώσει μόνο το μέλος. Η πολιτική μας ηγεσία και συμπεριλαμβάνω και εσά θα μας δώσουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε. Για το Brexit και τι ανησυχίε σχετικά πιστεύω πως έχουμε ε, καλύψει τα περισσότερα θέματα. Άκουσα και κάποιες ερωτήσεις για την ομόσπονδη υπηρεσία στις ΗΠΑ, την FAA και την αξιοπιστία των όσων κάνουν, όπως επίσης και η εξάρτησή τους από τον ε, κλάδο. Εγώ δεν έχω ελέγξει ούτε την FAA, ούτε τη δράση της, τουλάχιστον σχετικά με τα θέματα του ε, Boeing 737 ε, MAX. Ε, Έστησαν μια ομάδα εργασίας με μέλη διεθνείς εμπειρογνώμονες και νομίζω ότι έχουμε και Κινέζους ε, και Καναδούς και Ευρωπαίους στην ομάδα εργασίας που θα εξετάσει με επικριτικό πνεύμα το τι πήγε στραβά. Η έκθεση τους πρόκειται να δημοσιευθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, οπότε δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω τα πορίσματα, μια και σύντομα θα δημοσιευθεί. Το βέβαιο είναι πως όλες οι σχετικές αρχές και εμείς αντιμετώπιζαν με επικριτικό τρόπο αυτή την ανάθεση αρμοδιοτήτων για εγκρίσει από την FAA ε, προς την Boeing και είχαμε πει πιο συγκεκριμένο ότι αυτή η περίφημη δυνατότητα ε, ε, εμπλοκής ε, στις μανούβρες, αυτά τα ΕΜΑΚ που ε, θεωρούνται ότι προκάλεσαν σε μεγάλο βαθμό τα δύο δυστυχήματα, είχαν αυτοπιστοποιηθεί για να χρησιμοποιήσω το δικό σας όρο, κύριε Ρικέ, από την Boeing, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με το δικό μας σύστημα, που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτοπιστοποίηση. Γιατί αν συγκρίνουμε τα όσα κάνουμε εμείς με την FAA, εμείς έχουμε ένα σύστημα πολύ συγκεκριμένο, δομημένο, ε, με συγκεκριμένο τρόπο τη στιγμή της ανάθεσης αρμοδιοτήτων ε, στην ε, βιομηχανία τους. Εμείς είμαστε 800, δεν μπορούμε να ελέγχουμε κάθε γραμμή ε, προπολογισμού ή software που αναπτύσσει μια εταιρεία και είναι πολύ σημαντικό να συμφωνεί κανείς με τον ίδιο τον κλάδο πρώτον ποιες είναι οι μεθοδολογίες που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν και δεύτερον πώς γίνονται οι επαληθεύσεις σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά επίσης να γίνεται και μια συμφωνία για το οποιοδήποτε είναι καινοτόμο, οτιδήποτε είναι αυτοπιστοποιημένο, οτιδήποτε εμείς επιθυμούμε να εξετάσουμε, εξετάζεται από εμάς χωρίς να γίνεται ανάθεση και στις, με την Airbus και με τη Rolls Royce όποτε αρχίζει να τρέχει ένα καινούριο προϊόν διαπραγματευόμαστε μαζί τους για το ποια θα δούμε εμείς ως πρώτη προτεραιότητα και ποια όχι και ζητάμε να δούμε τα αποτελέσματα των δικών τους ελέγχων και μετά καταστρώνουμε τη γνώμη μας βασιζόμενοι στα όσα πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν, που είναι μια πολύ πιο λογική διαδικασία που την έχουμε στην Ευρώπη και κατά τη γνώμη μας λειτουργεί σωστά. Οπότε για την απάντηση που θέλω να σας δώσω κύριε Ρικέ και για κάποιους από συναδέλφους που ρώτησαν το ίδιο, ναι, είχε πρόβλημα, πιστεύουμε. Αυτή η σχέση ανάθησης αρμοδιοτήτων του ελέγχου ασφαλείας αυτών των MKA, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί περιμένουμε την έκθεση. Αυτό δεν θα είχε συμβεί στην, στο δικό μας σύστημα και μπορώ να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες αν το θέλετε. Και τώρα, και το σημαντικό για το πώς επηρεάζει το μέλλον και τη σχέση μας με την FAA, εδώ πρέπει να πω πως έχω πάρα πολύ σεβασμό για τους ομολόγους μου στην FAA για να απαντήσω στα όσα είπε ο κύριος Σκοτ γιατί το κατά πόσο υπηρετούν τον κλάδο ή τους πολίτες, όχι, τους πολίτες, αυτό το πιστεύω. Και μάλιστα, οι ηθικοί οι κανόνες που ακολουθούν είναι πραγματικά αυστηροί. Οπότε δεν έχω προβλήματα και δεν έχω αμφιβολίες καθόλου στο κατά πόσο είναι άξια αυτή η υπηρεσία. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι η μεθοδολογία τους και ενδεχομένως η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε εμείς όταν επικυρώνουμε, γιατί έτσι το λέμε, προϊόντα τα οποία έχουν επιστοποιηθεί από την FAA και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε και μαζί τους. Δεν μπορούμε να μπούμε αυτή τη στιγμή σε μια νέα περίοδο που θα κάνουμε συστηματική επαναπιστοποίηση όλων των σκαφών της Boeing γιατί θα κάνουν και αυτοί το ίδιο με εμά με την Airbus και όλους τους κινητήρες και όλα τα μικρά αεροσκάφη και νομίζω ότι αυτό είναι απλή επικάλυψη και δεν χρειάζεται ούτε μπορούμε. Πάντως έχουμε πάντα κατά νου τι συνέβη με τα δύο δυστυχήματα. Δεν έχω μια συγκεκριμένη απάντηση να σας δώσω, αλλά θα δούμε πώς θα συνεργαστούμε μελλοντικά. Για την κοινωνική διάσταση, Όντως, στο νέο βασικό κανονισμό, η ΆΣΑ, και αυτή είναι μια τροπολογία η οποία προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα εξετάζει και την κοινωνική διάσταση στον τομέα της, των αερομεταφορών για θέματα ασφάλειας. Δεν πρόκειται να κοιτάμε το μισθολογικό. Ξεκινήσαμε με μια πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου με τα συνδικάτα, με τους εργοδότες και ξεκινήσαμε επίσης να κάνουμε μια ε, να προετοιμάσουμε μια μεθοδολογία ε, ε, εξιολογικής, επιπτωσιολογική μελέτη, με συγχωρείτε, για να δούμε και την κοινωνική διάσταση. Οπότε, όπως κάνουμε την επιπτωσιολογική μελέτη για το περιβάλλον και την ασφάλεια, θα κάνουμε το αντίστοιχο και τα εργασιακά, έτσι ώστε μέσω της πλατφόρμας επίσης που έχουμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο εργαλεία, μεθοδολογία και πλατφόρμα και πρέπει να σας πω πως χαιρετίζω το διάλογο που κάνουμε μέσω αυτών και έχουμε μια ακόμα καινοτομία μέσω του βασικού κανονισμού ε, και οι αποσκευές. Ξέρουμε πως το θέμα ε, του handling είναι κοινωνικά πολύ ευαίσθητο και πιστεύω πως στο συζήτηση που ξεκινήσαμε με τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα προχωρήσουμε σε ένα θέμα ε, σημαντικό για την ασφάλεια με το όλο θέμα τους, ε, της διαχείρισης των ε, αποσκευών έτσι ώστε να καλύψουμε και εκείνο τον τομέα. για την περιβαλλοντολογική διάσταση, έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε κάτι το οποίο ε, ρηπαίνει με κάτι το οποίο επίσης είναι βλαβερό για τον πλανήτη. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και δεν πιστεύουμε πως η ηλεκτρική ενέργεια είναι και η μοναδική απόκριση που μπορούμε να δώσουμε. Γιατί κάποιος από σας είπε πως έχουμε προβλήματα με τους ορευτές ενέργειες και έχουμε επίσης και με την ισχύ των ηλεκτρικών κινητήρων, γιατί μιλάμε για μεγάλα αεροσκάφη. Οπότε δεν πιστεύουμε που σε τούτη εδώ τη φάση, και όταν λέω εμείς, δεν πιστεύουμε, νομίζω αυτό καλύπτει και την σχετική βιομηχανία, πως η ηλεκτρική ενέργεια είναι η πανάκια που θα λύσει τα θέματα αυτά στις αεροπορικές μεταφορές. Για τους θερμικούς κινητήρες ενδεχομένως, ναι, μπορεί να τους αντεκαταστήσει στα μικρότερα σκάφη, αλλά όχι για τα επιβατηγά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε εναλλακτικής ε, ε, λύσεις για την προώθηση, ίσως ε, ε κύτταρα, είτε για προώθηση μέσω λοιπόν ε, κυτάρων υδρογόνου, είτε κάτι εναλλακτικό. Είμαστε ανοιχτοί και θα ακούσουμε ό,τι έχουν να μας πούν τα ερευνητικά κέντρα, ο κλάδος, εσείς. Ο ρόλος μας για το περιβάλλον είναι να συντάξουμε τα πρότυπα και να πιστοποιούμε τους κινητήρες των ε, αεροσκαφών σε σχέση με τα πρότυπα αυτά. Και είναι σε ε, καπνό, σε σωματίδια, σε διοξίδιο του άνθρακα, σε διοξίδιο του θείου και σε ηχορύπανση τα πρότυπα τα οποία έχουμε και αυτά εφαρμόζουμε. Αυτά είναι τα εργαλεία που έχουμε και για οποιοδήποτε νέο προϊόν μπορούμε να πούμε αν ανταποκρίνεται στα πρότυπα αυτά ή όχι. Ένα από τα όρια που έχουμε είναι πως όλα τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να είναι παγκόσμια πρότυπα. Γιατί οι κινητήρες προέρχονται για παράδειγμα από τη ΣΥΠΑ ή το αντίστροφο, τα σκάφη από τα, τη ΣΥΠΑ κτλ. Τι σημαίνει αυτό χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εγκρίνουμε πιο περιοριστικά όρια, αλλά νομίζω ότι η φωνή μας ακούγεται, αλλά χρειάζεται χρόνο. Και είναι και μία... Είναι και ένα έμισο εργαλείο για φορολογία δεν μπορούμε να επιβάλλουμε. Να απαγορεύσουμε ε, προσγειώσεις και απογειώσεις δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε είναι ένα έμεσο εργαλείο υπέρ του περιβάλλοντος, το οποίο με οδηγεί ε, στις ερωτήσεις για την ηχορύπανση. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, θα αποτελέσει βασική πρόκληση στο μέλλον. Και για το λόγο αυτό δίνουμε αυτή τη τεράστια μάχη κατά του σχεδίου για τα υπερχητικά αεροπλάνα όχι για κάποιο πρόβλημα με τα σκάφη αυτά, αλλά θα λέμε, λέμε πως οποιοδήποτε υπερηχητικό jet ε, που θα απογειώνεται από ευρωπαϊκό αεροδρόμιο θα πρέπει να απογειώνεται κάνοντας λιγότερο θόρυβο από ότι ένα συμβατικό. Γιατί σήμερα τα μοναδικά πρότυπα που έχουμε είναι αυτά ε, που ισχύαν για το Concorde, το οποίο όταν απογειωνόταν, πρέπει να σας ε, το πω, ε, κατανάλωνε όλη την ηχητική δυνατότητα της συγκεκριμένης ημέρας. Άρα λοιπόν ξέρω πως θα με στηρίξετε, θα είναι πολύ δύσκολη η μάχη κατά τον είπα στο σημείο αυτών που έχουν πέντε σχέδια για υπηρεχητικά σκάφη στη ΗΠΑ, τα οποία παρακολουθεί στενά ο Λευκός Οίκος. Και αυτή τη στιγμή η Αμερικανική διοίκηση τους προωθεί και θέλουν να έχουν ε, πρότυπα διεθνή για τις απογειώσεις των επιχειρητικών που είναι πολύ ψηλότερα από αυτά που έχουμε για τα σημερινά συμβατικά αεροσκάφη και δεν νομίζω ότι το επιθυμούμε αυτό στην Ευρώπη. Για, την, ε, για το οικολογικό σήμα δουλεύουμε πάνω στο θέμα αυτό και αυτό που έχουμε υποέλεγχο είναι για τα νέα σκάφη είναι οι εκπομπές ήχων, οι εκπομπές διεξιδίων, σωματίδιο κτλ. Και πρέπει να σας πω πως εκεί είναι εύκολο να λύσουμε το θέμα του σήματος. Όλα αυτά έχουν δημοσιευθεί και ελπίζουμε και πριν τα τέλη της χρονιάς να τα έχετε. Είναι πολύ πιο περίπλοκο για τα αεροσκάφη, για τις αεροπορικές εταιρείες, Εκεί ξεκινήσαμε κάποιες προσπάθειες και με τα αεροδρόμια και με τις αεροπορικές εταιρείες για το τι ακριβώς θέλουμε να συμπεριλάβουμε σε αυτό το σήμα. Τη λειτουργία μόνο του σκάφους ή θέλουμε να συμπεριλάβουμε και την ανακύκλωση, για παράδειγμα, των υλικών και τέτοιου είδους ζητήματα. Όλα τα θέματα ακόμα είναι ανοιχτά. Ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε σε τεχνικό επίπεδο τις παραμέτρους που πρέπει να λάβουμε υπόψη, γνωρίζοντας ότι οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να είναι σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και απόλυτα ε, ελέγξιμο από ΜΚΟ ή οποιονδήποτε θέλει να εξετάσει τις παραμέτρους και τη μεθοδολογία υπολογισμού που ακολουθούμε. Είναι όλα λοιπόν ανοιχτά. Δώσαμε ένα χρόνο προθεσμία για να καταλήξουμε σε πρόταση και ελπίζω πως θα με καλέσετε να σας την παρουσιάσω όταν φτάσει και νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και για τους πολίτες και για τους επιβάτες. Για τα μη επανδρομένα ε, αεροσκάφη και για τα αεροταξί μας ρωτήσατε αν έχουμε καθυστερήσει ή όχι σε σχέση με άλλα κράτη. Νομίζω ότι εμείς είμαστε πολύ μπροστά εάν συγκρίνουμε με τους υπόλοιπου, γιατί το πιο εξελιγμένο, τα πιο εξελιγμένα σχέδια ε, για αεροταξί είναι στην Ευρώπη δύο γερμανικές εταιρείες οι οποίες νομίζω σε επίπεδο τεχνικής ορίμανσης είναι πιο μπροστά και υπάρχει μία χώρα την οποία γνωρίζω που είναι μπροστά από μας για την εμπορική χρήση ε, drones για την παράδοση εμπορικών αγαθών σε ε, αστικές περιοχές είναι η Αυστραλία η οποία ε, λειτουργεί ένα project της Google Wings που στην Καμπέρα τα τελευταία δύο χρόνια παραδίδει πακέτα και στις συζητήσεις που κάναμε μαζί τους προσπαθήσαμε να συζητήσουμε το τι γίνεται. Αυτά τα μη επανδρομένα σκάφη των drones είναι κάτι το οποίο λειτουργεί σε πολύ τοπικό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχει παγκόσμια πρότυπα για ό,τι έχει να κάνει με τα σκάφη αυτά. Αλλά προσπαθήσαμε να μοιραστούμε ευέλικτε πρακτικέ και εμπειρίε και οι Αυστραλοί. Ομόλογοι μα είπαν πω. το feedback που έλαβε από τους πολίτες της ε, Καμπέρας δεν είναι ότι φοβούνται ότι θα τους πέσει κάτι στο κεφάλι, είναι ο θόρυβος. Γιατί είναι πολύ θορυβόδη. Οπότε, εάν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός και νομίζω ότι το θέλουμε, η χρήση των drones στις πόλεις δημιουργεί δύο μεγάλα ζητήματα και εκεί εμείς χρειάζεται να λάβουμε και μία απόκριση από την κοινωνία. Πρώτον, ποιο είναι το επίπεδο ασφαλείας που θέλουμε, πόσο κίνδυνο μπορούμε να δεχτούμε και οποιοδήποτε πολύς περπατάει στον δρόμο, σε ποιο βαθμό θέλει να είναι εκτεθειμένο σε ντρόν που πετάει πάνω από το κεφάλι του. Αυτό είναι το πρώτο. Έχω την απάντηση, αλλά δεν ξέρω αν θα δώσετε και εσείς την ίδια. Και το δεύτερο, ποιο είναι το αποδεκτό επίπεδο ηχορύφανσης για τις πόλεις μας. Και κυρία Ντέλη, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν, γιατί όλα αυτά θα ενεργοποιήσουν πάρα πολλούς περιορισμούς στον τρόπο που θα εξελιχθούν, ε, εξελιχθεί ο κλάδος των μη επανδρομένων σκαφών και κυρίως ε, το θέμα του ήχου, γιατί αυτή τη στιγμή τα αποδεκτά όρια είναι τόσο χαμηλά που κανένα από αυτά που είναι στην παραγωγή δεν μπορούν να υπερίπτανται πάνω από τις πόλεις μας. Ε, για παράδειγμα, ε, μπορούν να πετάνε μόνο πάνω από ποτάμια κτλ. Και βέβαια, αν βάλουμε κάποιες μεγαλύτερες απαιτήσει ασφάλειας, μπορεί να ε, αυξηθεί πάρα πολύ το βάρος αυτών των σκαφών, των αεροσκαφών. Για τα θέματα του κυβερνοχώρου. Έχουμε αυξήσει τους πόρους μας. Ε, δεν είναι βέβαια πολύ εύκολο να βρει κανείς ε, κατάλληλο δυναμικό και είναι πολύ ακριβό. Έχουμε προσλάβει όμως τρεις εμπειρογνώμονες, αναγνωριμένους εμπειρογνώμονες ε, στην κυβερνοαεροπορία και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό. Χρειαζόμαστε περισσότερους σπόρους, διότι αυτό το θέμα γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Αναγνωρίζουμε ότι η αδυναμία της αεροπορίας ε, στην κυβερνοασφάλεια είναι η αδυναμία του συνόλου της αλυσίδιας προμήθειας. Μπορεί ε, η Boeing ή η Airbus να παραδίδει αεροπλάνο απόλυτα κυβερνοασφαλές, το οποίο όμως θα έχει ζωή 30 ετών. Και πολλές διαφορετικές εταιρείες θα εγκαταστήσουν νέο λογισμικό, θα το συντηρήσουν κλπ. Και από εκεί προέρχεται ο κίνδυνος. Καθώς και για την ε, κατάρτιση των πιλότων, ε, των ε, μηχανικών κλπ. Πρέπει δηλαδή, να φροντίσουμε καθόλου τη διάρκεια της αλυσίδας προμήθειας να διασφαλίζουμε την κυβερνοασφάλεια. Και αυτό προτείνουμε να γίνει με νέο κανονισμό, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί του χρόνου. και με τα θέματα κυβερνοασφάλειας συνδέεται και η ψηφιοποίηση, η προστασία των δεδομένων, ε, τι είδους δεδομένα χρησιμοποιούμε. Είμαστε αρκετά τυχεροί στον τομέα μας, ε, διότι χειριζόμαστε ε, τεχνικής φύσης δεδομένα. Αλλά, για παράδειγμα, έχουμε αρχίσει την εφαρμογή ενός μεγάλου ψηφιακού προγράμματος όπου συγκεντρώνουμε δεδομένα από όλες τις στήσεις της Ευρώπης ε, και έχουμε πετύχει συμφωνία με ε, τις οργανώσεις πιλωτών για να γνωρίζουμε τι ακριβώς κάνουμε, ε, ποια ε, δεδομένα θα πρέπει να ανωνυμοποιούνται κλπ. Επίσης, πράγματι έχουμε ενημερωθεί για το θέμα για το ε, ατύχημα του αεροπλάνου με τον ε, έναν κινητήρα. Είναι ένα από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Ήδη έχουμε εντοπίσει κάποιες από τις αιτίες των προβλημάτων και το παρακολουθούμε αυτό πολύ στενά, διότι αυτό το περιστατικό με το 330 είναι ένα θέμα που παρακολουθούμε στενά. Όσον αφορά το θέμα της Smart Wings, η οδηγία προς τους πιλότους σε όλο τον κόσμο δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την Ευρώπη, είναι το πλήρωμα να προσγειωθεί στο πλησιέστερο κατάλληλο αεροδρόμιο. Το πλήρωμα δηλαδή αποφασίζει τι, ποιο είναι κατάλληλο και αυτό έχει να κάνει με το βάρος του αεροσκάφους, ε, του, τον καιρό, έχει να κάνει με το μήκος του διαδρόμου προσγείωσης ε, κλπ. Ζητάμε από τα αεροπλάνα να προσγειωθούν το συντομότερο δυνατό όταν υπάρχει ένα θέμα ασφάλεια, όταν έχει πάρει φωτιά ένα κινητήρα, για παράδειγμα. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση, όπου είναι υποέλεγχο το πρόβλημα, η οδηγία σε όλο τον κόσμο είναι προσγείωση στο πλησιέστερο ε, κατάλληλο αεροδρόμιο. Έτσι λοιπόν η απόφαση να στο πλήρωμα. Ξέχασα κάτι το χρονοδιάγραμμα για την απογείωση των Boeing Max. Αυτό είναι ένα θέμα ανοιχτό. Κατά τη συζήτηση με την FAA τον Απρίλιο μας είπαν ότι τον Μάιο ήδη θα ξαναπετάξουν τα αεροπλάνα αυτά. Ε, στη συνέχεια είχαμε συνέχεια καθυστέρηση ενός μήνα. Βέβαια, καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να σα δώσω χρονοδιάγραμμα, διότι θέλουμε να είμαστε σωστοί, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάρτιση, πράγματι. Θεωρητικά μπορεί να έχει, έχει άλλες απαιτήσει ο ΕΑΣΑ και άλλες Ηνωμένε Πολιτείε. Κάνουμε όμως ότι μπορούμε να μην υπάρξει μια τέτοια κατάσταση, διότι αυτό δεν θα έχει νόημα σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή να χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση στην Ευρώπη από ό,τι στις ΗΠΑ ή σε άλλα μέρη του κόσμου. Και τέλος, όσον αφορά τη διεθνή κοινότητα και την φήμη, το, το γόητρο του FAA, πρέπει να πω ότι το FAA βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. διότι όταν πούν ότι ωραία εντάξει προχωράμε, είναι πάρα πολύ πιθανό εθνικές αρχές να θέλουν και μια δεύτερη γνώμη ή τρίτη γνώμη. Και κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε πριν ένα χρόνο. Νομίζω ότι θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τη διεθνή ιεραρχία ή τη σχέση ανάμεσα στις διάφορες ε, αρχές. Έκανα ό,τι μπορούσα για να απαντήσω. Ε, παρακαλώ, μη διστάσετε να έρθετε απευθεία σε επαφή μαζί μου αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις. Υπάρχει κάποιος που έχει να κάνει μια παρατήρηση, μια άλλη ερώτηση. Πολύ γρήγορα σας παρακαλώ, έχουμε μόνο 7 λεπτά. Παρακαλώ. Θα ήθελα να συνεχίσω την ερώτηση που έκανα για το Brexit. Δηλαδή, αν τελικά η Μεγάλη Βρετανία ε, φύγει, το Ηνωμένο Βασίλειο φύγει στις 31 Οκτωβρίου χωρίς συμφωνία, τι θα γίνει όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο την 31η Οκτωβρίου. Ε, νομίζω ότι ανησυχούν οι πολίτες στην πατρίδα μου. Γιατί, ναι, θα γίνουμε τρίτη χώρα. Και τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Ποια είναι, λοιπόν, τα πρακτικά βήματα που θα πρέπει να κάνουμε. Ποιε οι διασφαλίσει που μπορούμε να δώσουμε στους επιβάτε όσον αφορά την ασφάλειά τους. ούτω ώστε να εξακολουθούν να είναι συμβατά με αυτά που υπάρχουν και την 31η Οκτωβρίου. Μια τελευταία ερώτηση, σας παρακαλώ πολύ γρήγορα. Δεν απαντήσατε όσον αφορά την δική σας μελέτη για την αποτελεσματικότητα ε, του περιορισμού του χρόνου πτήσης ε, και των νυχτερινών πτήσεων. Και επίσης όσον αφορά την διαδικασία επικύρωσης, ο ΕΑΣΑ έπαιξε ρόλο ε, όσον αφορά τα Boeing 737 το 2016 ε, είχατε εντοπίσει το πρόβλημα για το οποίο, το οποίο είναι, ε, ήταν η αιτία αυτών των δυστυχημάτων, αλλά δεν μπορούσατε να εφαρμόσετε τα μέτρα. Τι θα κάνετε λοιπόν ε, στο μέλλον. Όσον αφορά το Brexit. Το θέμα λοιπόν είναι, όπως είπαμε, η ασφάλεια. Το τονίζουμε υπάρχουν τρίτες χώρες για τις οποίες το επίπεδο ασφάλειας για τους επιβάτες είναι τόσο υψηλό, αν όχι πιο υψηλό, ε, από ε, το ευρωπαϊκό. Η Σιγκαπούρη, για παράδειγμα. Όταν μιλάμε για τρίτη χώρα, Λοιπόν, δεν σημαίνει αυτόματα ότι μιλάμε για χαμηλότερα πρότυπα ασφαλεία. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση όσον αφορά λοιπόν την ασφάλεια, και αυτό ισχύει για όλα τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα υψηλότερα. Και βέβαια, όταν έχετε τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας, ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα δεν θα πέστε στα κατώτερα, στα χαμηλότερα. Νομίζω λοιπόν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να έχει πολύ αυστηρά ε, πρότυπα ασφαλείας. το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη σήμερα τηρεί πλήρω την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο βεβαίω θα υπάρχουν οπωσδήποτε κάποιε διαφορές ανάμεσα στην νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και την ενωσιακή. Και αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι ότι δεν θα είμαστε πλέον εκεί για να ελέγχουμε τι γίνεται. Πρέπει λοιπόν να βρούμε πώ μπορούμε στη συνέχεια να συνεργαστούμε. Και όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Ντάλι, συζητήσαμε με πολλά σωματεία ε, για τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Εντοπίσαμε λοιπόν κάποια προβλήματα, αλλά υπάρχουν και θέματα που δεν έχουν προβλήματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι, αυτή είναι η πρώτη φάση λοιπόν τη της μελέτης η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για το μέλλον. Δεν πρόκειται βεβαίως να ε, δούμε όλο το σύνολο της νομοθεσίας, αλλά θα πρέπει να δούμε ε, σε κοινωνικό επίπεδο ποιοι θα είναι οι συνομιλητές μας για να μπορέσουμε να πάμε πιο πέρα. Και πρέπει, μπορώ μάλλον να σας εγγυηθώ, ότι όσον αφορά την ε, κατάρτιση και όσον αφορά την ε, επαναλειτουργία των Boeing 737 θα κάνουμε τα απαραίτητα. Ευχαριστώ πολύ Κυριακή. Μία τελευταία παρατήρηση όσον αφορά το κοινωνικό σκέλος. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας στείλει λοιπόν το περίφημο πακέτο για την αεροπλοεία και να έχουμε λοιπόν και το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό σκέλος. Το δεύτερο είναι ότι ναι, ε, εσείς ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός δεν έχετε τη δυνατότητα να θεσπίσετε κοινωνικά ε, πρότυπα. Σας ευχαριστούμε πολύ Κυριακή. Ε, χαρήκαμε ιδιαίτερα που σας είχαμε κοντά μας, όπως πάντα. Ε, μας παρέχετε συχνά πληροφόρηση και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία στο μέλλον και θα έρθουμε να σας δούμε μάλιστα. Είστε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας και είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι όλα αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια, με το Brexit, με το περιβάλλον, με το μέλλον του κλάδου, δεν το είπαμε αρκετά, αλλά ο διεθνής ανταγωνισμός για τον κλάδο αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ε, αυξημένος και αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά, λοιπόν, θα πρέπει να τα ξαναδούμε πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε και σας χειροκροτούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνουμε εδώ. Να σας πω ότι οι επόμενες συνεδριάσεις μας, οι επόμενες συνεδριάσεις θα είναι στις 23 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Τέλος συνεδρίασης.